κοιτή της, αυτής από την κυρία Γέννησεν η οποία δεν επανεξελέγει. Θα ήθελα λοιπόν να την ευχαριστήσω ακόμα και αν δεν βρίσκεται εδώ σήμερα και να ευχαριστήσω πολύ και την Σαβελίνα από τη Γραμματεία η οποία έκανε εξαιρετικό προπαρασκευαστικό έργο. Τώρα, καταρχάς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει στεναρά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και πιστεύει ότι είναι αναγκαίο η Ένωση να βελτιώσει περαιτέρω την εποπτεία σε ενωσιακό επίπεδο. Οι αρχές ιδρύθηκαν το 2011 εν μέσω της οικονομικής κρίσης όπου και ανέλαβαν καθήκοντα από τις προηγούμενες αρμόδιες επιτροπές. Είναι, πιστεύω, ο ακρογωνιαίος λίθος μιας, ε, σωστά, μιας ε, σωστής ε, χρηματοοικονομική αγορά και συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση καθώ και στην αποφυγή νέων κρίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Με ανησυχεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι υπάρχει, υπάρχουν πολύ μειωμένα, μειωμένα κονδύλια για τον προϋπολογισμό του 2015. Και προτείνουμε μια και όλες οι εποπτικές αρχές ε, δεν έχουν αρκετό προσωπικό να διατηρηθεί ο αριθμός των ε, μέχρι τώρα υπαλλήλων. Μετά από συζητήσεις και δικές μου και των, της γραμματείας με τις αρμόδιες αρχές ε, τα επιχειρήματά τους μας φάνηκαν αρκετά πιστικά και η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ίδια άποψη. Προτείνω λοιπόν να επαναφέρουμε τους ε, αριθμούς που ε, προτείνει και η Γαμαδέλτα ΜΑΡΚΤ. Και ο λόγος της επαναφοράς αυτών των ε, κονδυλίων είναι προφανής. Τα τελευταία δύο χρόνια οι τρεις αυτές εποπτικές αρχές ανέλαβαν αυξημένα καθήκοντα συμπεριλαμβανομένης της ε, παρακολούθησης, της εφαρμογής και της συμμόρφωσης της νομοθεσίας. Επίσης, ανέλαβαν καθήκοντα που απορρέουν από την ε, ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης και για το λόγο αυτό θα χρειαστούν επιπλέον μέσα προπολογισμού για να μπορούν να εκπληρώσουν τον εποπτικό του ρόλο όπως αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό για τις εποπτικές αρχές. Είναι επίσης σημαντικό οι αρχές αυτές να έχουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε να μπορέσουν να ε, πληρώσουν ικανοποιητικά το έργο τους. Και συνήθως δεν εγκρίνω μια λευκή επιταγή, ούτε εδώ ούτε και στην πατρίδα μου, εάν αυτές δεν είναι εμπεριστατωμένες και στηριγμένες με επιχειρήματα. Αλλά σε μια συζήτηση με τον ε, αντικαταστάτη του Επιτρόπου κυρίου Λεβαντόφσκι μας ε, παρουσιάστηκε η κατάσταση του προϋπολογισμού. Όμως, εάν δεν υπάρχει στήριξη από τον ε, προϋπολογισμό, τότε δεν, μπορούμε, δεν μπορούν οι υποπτικές αρχές να κάνουν και το έργο για το οποίο έχουν προβλεφθεί. Και αυτό αφορά και την απασχόληση υπαλλήλων οι οποίοι δεν είναι σε ε, πολλές περιπτώσεις και οι πλέον αρμόδιοι για τα καθήκοντά τους. Και δεν μπορούν λοιπόν να φέρουν σε πέρας τις εργασίες οι οποίες τους έχουν ανατεθεί. Επίσης, ε, πιστεύουμε πως οι ισχύουσες διευθυντήσεις χρηματοδότησης βασίζονται σε ένα μικρό σύστημα, μεικτό σύστημα χρηματοδότησης και αυτό δεν είναι ευέλικτο. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να προτείνουμε μέχρι το 2007 να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό σύστημα που να βασίζεται σε καταβολή τελών από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Θα χαρώ λοιπόν να συζητήσουμε την γνωμοδότηση αυτή με τους κοιόδες ηγητές και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ευχαριστώ δίνω το λόγο στους σκιώδεις ηγητές από τις πολιτικές ομάδες. Η Ιβάνα Μάλετης για το ΕΛΚ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόρβαλτς. Νομίζω ότι έχετε εξηγήσει πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει εμείς να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για αυτές τις τρεις σημαντικές εποπτικές αρχές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε σωστή εφαρμογή και ομοιόμορφη ε, εφαρμογή όλων των κανόνων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς αυτή την ε, ομοιόμορφη εφαρμογή θα χάσουμε τα δυνητικά ωφέλη μιας κοινή εποπτικής αρχής για αυτές τις τρεις αρχές, για αυτούς τους τρεις φορείς. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τον αριθμό του, των μελών του προσωπικού τους και τον προϋπολογισμό τους. Αυτά περιλαμβάνει η πρόταση με την οποία συμφωνούμε. Αυτό το οποίο πρέπει να, να λάβουν υπόψη αυτές οι τρεις αρχές είναι αν αυξήσουν πολύ τον αριθμό του προσωπικού τους θα πρέπει να αναζητήσουν πιο πεπειραμένο προσωπικό διότι αν το προσωπικό τους δεν είναι πεπειραμένο μπορεί να έχουν δυσκολίες. Χρειάζονται πολύ επαγγελματικό προσωπικό και τον κατάλληλο προπολογισμό για να το προσλάβουν Αυτά λοιπόν από την πλευρά του ΕΛΚ θα θέλαμε να παρατηρήσουμε προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούντβιξον για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το θαυμάσιο σχέδιο έκθεσής του και ευχαριστώ επίσης για τις ε, λογικές προτάσεις που έχει διατυπώσει σε επίπεδο ποσών για τον προϋπολογισμό νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τα θεμελιώδη στοιχεία αυτής της έκθεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο των εποπτικών αρχών. Αυτό ήταν φυσικά ως Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων η πρώτη μας προτεραιότητα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια δύσκολα, λεπτά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τρεις αυτές εποπτικές αρχές βλέπουν να αυξάνεται συνέχεια ο φόρτος εργασίας τους λόγω του μεγαλύτερου όγκου νομοθεσίας που εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτό είναι σημαντικό για μας να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Ο κίνδυνος περιορισμένης ή ελλειπούς εφαρμογής των κανόνων αυτών από αυτές τις αρχές εξακολουθεί να υπάρχει. Αν δεν είναι, αν είναι αποδυναμωμένοι αυτοί οι φορείς δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν σωστά την εποπτική τους λειτουργία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η μεταρρύθμιση η οποία είναι απαραίτητη και να υπάρξει και ο έλεγχος της εφαρμογής αυτής της μεταρρύθμισης. Η Κομισιόν έχει μια σχετικά αρνητική αντιμετώπιση γιατί για το 2015 προτείνει ή να μειώσει ή στην καλύτερη περίπτωση να κρατήσει σταθερή τη χρηματοδότηση για τους τρεις αυτούς φορείς. Χρειάζονται περισσότερο περιθώριο λιγμών για τους ε, φορείς αυτούς, κάτι όμως που δεν δέχεται η Κομισιόν και δεν καταλαβαίνω γιατί. Θα έπρεπε να ενισχύσει τις, ε, τους τρεις αυτούς ε, φορείς και ενώ τους δίνει περισσότερη εργασία δεν τους δίνει τους απαραίτητους πόρους. <clears throat> Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη χρηματοδότηση και αυτά τα οποία προτείνει ο κύριος Τόρβαλτ είναι απόλυτα λογικά και έχουν ένα εξισορροπημένο χαρακτήρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να δεχτούμε τα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται στην έκθεση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δεχτούμε όλες αυτές τις λεπτομεριακές ε, αναγραφές στοιχείων, αλλά θα πρέπει να έχουν τους απαραίτητους πόρους αυτές οι τρεις αρχές και φυσικά θα πρέπει να σκεφτούν και για τις δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης στο μέλλον από εισπατώμενα τέλη. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να απορροφούν λιγότερους πόρους ώστε να αποδίδονται περισσότεροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή θα πρέπει η Κομισιόν να βρει την κατάλληλη λύση και να δημιουργήσει την κατάλληλη σχέση και το κατάλληλο κλίμα μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών ε, εποπτικών αρχών. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η αυτοχρηματοδότηση αυτών των ε, φορέων. Θα ήταν πολύ χρήσιμο όμως να ξέρουμε κατά πόσο είναι δυνατό να έχουμε χρηματοδότηση και από το χρηματοπιστωτικό τομέα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν παράλληλα μερικά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να θέσουμε. Με το πρόγραμμα Φισκάλης 2020 και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να λειτουργήσουν για να υπάρξει καλύτερη υποπτία. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να ληφθεί η απαραίτητη μέρημνα. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να βρεθούν έξω από τους φορείς αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κέιτ. Σας ευχαριστώ. Όπως και σήμερα το πρωί. Ελπίζω η έκθεση αυτή ε, θα περάσει από σε ένα σκιώδη συγγητή το ταχύτερο δυνατόν. Θα ήθελα να πω ότι ιστορικά η ομάδα μας έχει υποστηρίξει τον συντονιστικό ρόλο τον οποίο παίζουν ε, οι αρχές αυτές εποπτείας. Υποστηρίζουμε επίσης και τη σωστή τους λειτουργία και τον τρόπο υποστηρίξαμε με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Πριν φτάσουμε στην, θα έλεγα, στην ενδιάμεση, στον ενδιάμεσο ανασχεδιασμό, θα πρέπει να δούμε τι ανάγκες έχουν σε οικονομικό επίπεδο, ποιος θα πρέπει να είναι ο προϋπολογισμός τους. Να δούμε τι σωστότερες προτεραιότητες μπορούμε να βάλουμε μέσα σε αυτό τον προϋπολογισμό. Είναι σαφές ότι αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι αρχές δεν έχουν εξοδεύσει περισσότερα από όσα θα έπρεπε και γι' αυτό πρέπει να τις βοηθήσουμε. Έχουν βέβαια ένα όριο η ΕΣΑ. Εξαρτώνται εν πολλής από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακόμα περισσότερο αυτούς τους, εθνικούς, ε, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που υπάρχει βεβαρημένη ατζέντα για τη λειτουργία τους το πιο περιοριστικό θα έλεγα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό είναι το θέμα των πόρων. Και πολύ συχνά οι εμπειρογνώμονες κάθονται στα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε λοιπόν να ε, ε, διευκολύνουμε την κατάσταση τη δύσκολη στα δημοσιονομικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες τουλάχιστον κατά 25% του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να βοηθήσουμε και οι εθνικές αρχές ε, να ε, χρησιμοποιήσουν σωστά ε, τον, το, αυτό το συγκεκριμένο εγχειρίδιο των κοινών κανόνων το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις εργασίες των εποπτικών αρχών. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός και το εκτιμούμε, αλλά θα αλλάξει αυτό και δεν θα είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε την ευελιξία τους. Ο εισηγητής έχει αναφερθεί και στα προβλήματα που έχουν οι αρχές αυτές σε επίπεδο πρόσληψης. Όταν εμείς δημιουργήσαμε τα ΕΣΑΣ είπαμε ότι το πρόβλημα το γλωσσικό είναι σοβαρό πρόβλημα και θα συνεχίσει να είναι. Υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν μια δεύτερη γλώσσα. Αν θέλουμε λοιπόν να επιβάλλουμε τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ΕΣΑ, δηλαδή στις αρχές αυτές, είναι λάθος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσλαμβάνει εμπειρογνώμονες, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες για το ποιοτικό προσωπικό το οποίο αυτή τη στιγμή ε, διεκδικούν και το ίδιο συμβαίνει επίσης και με υπηρεσίες όπως ε, οι αρχές αξιολόγησης, οι εξωτερικές υπηρεσίες αρχαιολόγησης κτλ. Η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι πάντως πρώιμη και θα πρέπει όταν αναθεωρήσουμε γενικά τη λειτουργία των ίσα, όταν έρθει η στιγμή αυτή να δούμε τι θα κάνουμε. Η ανεξαρτησία τώρα των αρχών αυτών, από τι είναι ανεξάρτητες ή από τι πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Ε, θέλω να είναι και εκεί ανεξάρτητες, θέλω να είναι ανεξάρτητες και στις στάσεις που δίνουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια ανάληψη ευθύνη από τα διοικητικά του συμβούλια. Λοιπόν, η λέξη ανεξαρτησία σημαίνει πολλά σε πολλούς και πολλές φορές διαφορετικά. Και υπάρχει κι άλλο ένα μικρό θέμα εδώ. Η ευελιξία θα πρέπει να αυξηθεί. Μπορεί να γίνει στα πλαίσια του παρόντος προϋπολογισμού και νομίζω ότι πολλοί φίλοι από άλλες πολιτικές ομάδες θα με βοηθήσουν να διασφαλίσουμε την ευελιξία αυτών των αρχών εποπτείας που κάνουν μια τρομακτικά θετική δουλειά. Euh, euh, Σε σχέση με την έκθεση αυτή, Εξ ονόματος της ε, ομάδος μας θέλουμε να εκφράσουμε μια βασική επίκριση γιατί η έκθεση αυτή ακολουθεί μια ιδεολογική, γραμμή που είναι αντίθετη από τη δική μας εικόνα την, για την Ευρώπη. Είναι μια φεδεραλιστική, καπιταλιστική Ευρώπη όπου κυριαρχούν οι αγορές και που θεωρεί ότι οι νόμοι της αγοράς μπορούν να λύσουν τα προβλήματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και εμείς βλέπουμε από την ε, ιστορία ότι πρώτα οι νόμοι της αγοράς αστοχούν και όταν καταλάβουμε όλοι το αποτέλεσμα αυτής της ε, φιλελευθερωπής που οδηγεί σε καταστροφή, μόνο τότε γίνεται μια προσπάθεια κάπως να χαλιναγωγούνται οι νόμοι της ε, αγοράς. Το να γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια να αυξηθεί η ρύθμιση μετά από την κατάφορη απόδειξη της ε, αποτυχίας της αγοράς είναι ένα πολύ καλό δείγμα του λαθασμένου δρόμου που ακολουθεί η Ευρώπη. Γι' αυτό οι δικές μας επιφυλάξεις αφορούν κυρίως την ε, ανικανότητα των μηχανισμών της αγοράς να λύσουν τα προβλήματα αυτά, ιδίως όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι προϋπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνονται σταθερά και είναι φανερό ότι οι πόροι για να μπορέσουμε να προωθήσουμε μια μορφή εποπτείας που να είναι ελάχιστα αποτελεσματική κατά τη δική μας άποψη φυσικά δεν είναι παρόντες. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με την προφορική μου, με την προσωπική μου συγγνώμη άποψη ότι είμαι πλήρως πεπισμένος ότι η εποπτεία αυτή είναι σίγουρα από την μορφή αυτή υποπτήρηση είναι πολύ καλύτερα να έχουμε ένα κρατικοποιημένο χρηματοπιστωτικό τομέα από την κατάσταση που βλέπουμε τώρα είναι πολύ καλύτερο. Thank you. Sven Giegold, Greens. Ο Sven Giegold. Και εγώ προσβλέπω σε μια μακρά συζήτηση για τα θέματα αυτά. Αν συζητήσουμε τελικά για το αν θα πρέπει ο καπιταλισμός να έλθει σε ένα τέλος και να κοινωνικοποιηθούν όλες οι χρηματαγορές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αλλά εγώ θα ήθελα τώρα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή και να τον ευχαριστήσω για όλα αυτά που έκανε για τις επόπτικες αρχές. Θα με ενδιέφερε να ακούσω και από την Κομισιόν να μου εξηγήσουν γιατί θέλουν να περικόψουν τον προϋπολογισμό ενώ είναι φανερό ότι του χρόνου θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο μεγαλύτερος φόρτος εργασίας για αυτούς τους φορείς και θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν περαιτέρω και τα ίδια άκουσα και από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς. Στην αρχή δεν θέλανε αυτές τις περικοπές αλλά κατέληξαν σε μια τέτοια ρύθμιση. Αυτό είναι ένα διαρθωτικό πρόβλημα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και το έχουμε δει και σε προηγούμενε γνωμοδοτήσει για τον προπολογισμό στη δική μου από σε αυτήν του Βενελάγγεν, Πάντα υπάρχει αυτή η επιμονή να υπάρχει μια ανεξάρτητη γραμμή του προπολογισμού ώστε να μην υποχρεωμένη η Γενική Διευθύνση Μάρκτη Εσωτερικής Αγοράς να περικόπτει προϋπολογισμούς για να βοηθήσουν μια, ένα φορέα σε βάρος κάποιων άλλων. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε να αλλάξει η διάθεση του προϋπολογισμού ώστε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Και περαιτέρω εμείς υποστηρίζουμε το ότι <clears throat> οι εμπλεκόμενοι στην αγορά αυτοί δημιουργούν το κόστος αυτό και θα πρέπει σύμφωνα με τις θεωρίες του Πίγκο και αυτοί να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των ε, φορέων αυτών. Και θα θέλαμε επίσης να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει και μεγαλύτερη ε, γνώση και εμπειρογνωμοσύνη της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της ε, νομοθεσίας για τα χρηματοπιστωτικά θέματα, να έχουμε μια καλύτερη πολιτική επικοινωνία της Κομισιόν σε σχέση με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε αποκομίσει από προηγούμενους κύκλους διαβουλεύσεων για να δούμε αν υπάρχει πρόοδος για τα θέματα αυτά ή όχι και επιπλέον η χρηματοδότηση της ΕΦΡΑΚ και της ISB εξακολουθούν και στον τρέχοντα προϋπολογισμό και θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις Μάιστατ έχουν προχωρήσει όπως είχαμε συμφωνήσει όλοι και αν δεν έχουν προχωρήσει, αν δεν έχουν δοκιμήσει, θα πρέπει να σκεφτούμε αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες μας για τον τρέχοντα προϋπολογισμό για να τηρηθούν τα υπεσχημένα στον τομέα αυτό. Έχουμε παραδείγματος χάρη κάποια ερωτήματα σε σχέση με τους κανόνες IFRS και ISB αν έχουν σταματήσει να προωθούνται προς ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο εμείς δεν θέλουμε να συμβεί. Και λυπούμαστε για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να αποδυναμώσει τη Eurostat. Εμείς επιμείναμε εδώ και πολλά χρόνια να έχουμε μια ισχυρή υπηρεσία ευρωπαϊκών στατιστικών. Πιστεύουμε ότι ο αρχικός, η αρχική πρόταση της Κομισιόν για τον προπολογισμό της Eurostat θα πρέπει να επανέλθει και να μην υπάρξει μείωση. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πολύ. Αναλύσαμε την πρότασή σας και είδαμε ότι υπάρχει πρόβλημα και μία δυσαναλογία ανάμεσα στο προσωπικό ε, και στις διάφορες κατηγορίες του προσωπικού, τους βοηθούς, γραμματείς ε, και το, τα στελέχη, τα διοικητικά. Ιδιαίτερα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης ίσως ε, θα πρέπει να αποφύγουμε κάποιες απαράδεκτες μορφές ε, διοίκησης, αλλά ένα 20% επιπλέον είναι κάτι το, το πολύ λάθος. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση του προϋπολογισμού και θα πρέπει να υπάρξει μια ανακατάταξη των διαφορετικών κατηγοριών του προσωπικού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. θα... έχουμε μια γρήγορη διαδικασία του Catch the Eye και ο κύριος Μπάλτς έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ έχω την άποψη ότι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάπως ε, περίεργα. Έχω επικριτική στάση. Και πιστεύω ότι αυτά τα ποσοστά που αναφέρατε δεν μπορώ να τα δεχτώ. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ήμουν εισηγητής για το Omnibus 2. Και ήμουν υπεύθυνος και για... Ε, ε, και για ασφαλιστικά ζητήματα και επαγγελματικά ζητήματα. Και έχει δημιουργηθεί τώρα, έχουν δημιουργηθεί πρόσθετες αρμοδιότητες στις εποπτικές αρχές που σχετίζονται με αυτά. Τώρα, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον περιορισμένο προϋπολογισμό για να διεξάγει μελέτες και να συνεχίσει το έργο τότε πιστεύω ότι δεν θα το καταφέρει και εμείς εδώ δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Εγώ περιμένω μια βελτίωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά να πω ότι καλωσορίζω αυτήν την μικρή αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ερευνών. Σίγουρα είναι μια υπηρεσία η οποία είναι ωφέλιμη και στο μέλλον θα μπορέσει να ε, συνεισφέρει ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω αυτή την μικρή αύξηση, όπως είπα, των ε, κονδυλίων για την υπηρεσία αυτή. Όμως ε, πιστεύω πως δεν ήταν σωστή η κατανομή των πόρων. Κύριο Σόφιν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν στους ε, συμμετέχοντες ε, στην αγορά, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν. Βέβαια, ο αντίκτυπος ε, θα γίνει αισθητό στους, μικρούς, στους μικροκαταθέτες και στους μικροεπενδυτές στην Ευρώπη και όχι στους συμμετέχοντες στην αγορά. Χρειαζόμαστε ε, συστάσεις για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτά τα κονδύλια, διότι πρέπει να αποφύγουμε στο τέλος τα πράγματα να γίνονται όλο ένα και πιο ακριβά. Θα θέλαμε λοιπόν ε, να δούμε εάν όντω αυτό ο τομέα είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι θα γίνει με αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητά το λόγο. Τώρα λοιπόν θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, τον εκτελεστικό της Διευθυντή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαστε εδώ και οι τρεις και από τις τρεις εποπτικές αρχές και θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω εκ μέρους της ε, EBA, της δικής μου υπηρεσίας. Είναι μία από τις πρώτες επαφές ε, που έχω με το νέο κοινοβούλιο, η σημερινή, και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους κεώδης εισηγητές για τις ε, συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων που είχαν μαζί μας, γιατί αυτό μας βοήθησε να ε, δούμε περισσότερες λεπτομέρειες, να δούμε από πού προέρχονται τα αιτήματα του προπολογισμού και τι αυτά περιέχουν. Τώρα, θα ήθελα με λίγα λόγια να σας πω ότι από την σύσταση της EBA το 2011 και των υπόλοιπων εποπτικών αρχών, οι αρμοδιότητές μας αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε απόλυτη επίγνωση του ότι αυτή η αύξηση αρμοδιοτήτων δεν θα κρατήσει για πάντα και ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα εξισορροπήσουν τα πράγματα όμως, δυστυχώς δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η ώρα και προς το παρόν έχουμε μια επιθετική αύξηση αρμοδιοτήτων. Ο προϋπολογισμός μας βασίζονταν πάντα σε συγκεκριμένα αιτήματα, συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με λεπτομερείς αναλύσεις ε, και διάφορες μελέτες που καλούμαστε να κάνουμε. Και εμείς έχουμε απόλυτη διαφάνεια ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε πανέτοιμοι να σας δώσουμε κάθε εξήγηση και κάθε λεπτομέρεια που θα χρειαστείτε. Τώρα, ε, η νομοθεσία για την οδηγία IP είναι σχετικά πρόσφατη, όπως και η νομοθεσία για τον νέο μηχανισμό εξυγίανσης και το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Εμείς πρόσφατα λάβαμε μία νέα εντολή για το 2015 η οποία περιλαμβάνει 69 προϊόντα, τα οποία σχετίζονται με αυτή τη νέα νομοθεσία που μόλις ανέφερα. Δηλαδή 15 ρυθμιστικά πρότυπα που έχουν να κάνουν με την, με την εφαρμογή, τεχνικά πρότυπα, συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ως συμπληρωματικά ε, προϊόντα. Όλα, πιστεύουμε λοιπόν αυτά, δικαιολογούν το αίτημα που κάναμε για αύξηση του προϋπολογισμού μας και αύξηση του προσωπικού μας. Διότι πιστεύουμε πως ε, αυτό αντιστοιχεί στις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την στήριξη που μας δίνετε ως Επιτροπή ΕΚΟΝ και να σας πω ότι βρισκόμαστε στη διάθεσή σας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και να σας ε, κρατάμε ενήμερους για το τι κάνουμε και πώς ακριβώς το κάνουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Κάρλος Μοντάλπο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα και για την συνεχόμενη στήριξη που μας δίνετε. Φυσικά θέλουμε και εμείς και εσείς να Είμαστε επιτυχείς στο έργο μας. Τώρα θα προσπαθήσω να συνοψίσω το έργο μας και να στείλω και ένα μήνυμα στο τέλος. Καταρχάς, ο προϋπολογισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο προϋπολογισμός και ε, διοχετεύεται σε τέσσερις ε, τομείς. Ε, ακολουθούμε μια πολύ ειλικρινή προσέγγιση στο έργο μας ε, διάφανη και όπως ε, είπε και ο συνάδελφος και εμείς ε, θα είμαστε πρόθυμοι να καλέσουμε όποιον από εσάς επιθυμεί να έρθει και να δει πώς δουλεύει. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να εντοπίσουμε τους τομείς τους οποίους θέλουμε να εστιάσουμε και ο συνάδελφός μου στα δεξιά μου κάνει ακριβώς αυτό. Και τέλος ο προπολογισμό εγκρίνεται από του ευρωβουλευτές και έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες όπως γνωρίζετε. Τώρα στο αίτημα για τον προϋπολογισμό του 2015 έχει παρατηρηθεί μια αύξηση 3%. Όμως αν δείτε τα συστατικά στοιχεία αυτού του προϋπολογισμού θα δείτε ότι έχουμε περικόψει 12% του κόστου σχετικά με το 2014 και 13% σε σχέση με το 2013. Και ο μόνος τομέας στον οποίο ζητούμε αύξηση είναι ο τομέας του προσωπικού. Και αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ως υπηρεσία ότι έχουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις δικές σας και των Ευρωπαίων πολιτών, όμως ε, χρειαζόμαστε κονδύλια γι' αυτό. Τώρα, πώς καταρτίζεται ο προϋπολογισμός. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2013 για τις ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Και η προσέγγιση αυτή χωρίζεται σε τρεις ε, κατηγορίες στις ε, κατηγορίες που αρχίζουν μόλις, στις κατηγορίες που ήδη ε, υπήρχαν και στις, ε, και στα, στις νέες κατηγορίες, στα νέα καθήκοντα. Τώρα, στην πράξη όμως τι γίνεται. Για τον προϋπολογισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρει ακριβώς τα ίδια νούμερα του 2013 και τα έχει προσαρμόσει το 2015. Και για τις νέες αρμοδιότητες, Όμως και διότι φέτος η Δημοσιονομική Αρχή, εσείς δηλαδή και το Συμβούλιο, έλαβαν μία απόφαση να μας ε, δώσουν και έναν επιπλέον προϋπολογισμό. Και αυτές οι περικοπές του 10% που αναφέρατε σημαίνουν, με λίγα λόγια, ότι το ένα όργανο αγνοεί το άλλο. Το Συμβούλιο μας ζητά διάφορες εργασίες. Δεν τους ενδιαφέρει όμως ο προπολογισμό. Δεν θέλουν να ξέρουν πόσο κοστίζει όλο αυτό. Και μετά ερχόμαστε εδώ σε εσά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο, ε, μας στηρίζει, μας έχει ε, αναθέσει αρμοδιότητες, οι οποίες ολοένα και αυξάνονται. Μα στηρίζει όμως όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις, δηλαδή με την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γι' αυτό λοιπόν και με χαρά μου άκουσα τον εισηγητή, ο οποίος ανέφερε ότι θέλει να ε, επανεξεταστεί η πρόταση για τα κονδύλια που θα ε, διατεθούν. Και αυτό με χαροποιεί πολύ διότι πριν από δύο χρόνια έχουμε μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς ε, αυτό το θέμα. Και, υπός, και να σας πω και κάτι ε, προσωπικό. Όταν παντρεύτηκα, η γυναίκα μου μου είπε ότι η αγάπη δεν είναι μόνο λόγια, αλλά είναι και πράξεις. Και αυτό πόσο μεταφράζεται εδώ. Τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι μας λέει το Κοινοβούλιο. Αν ακούγαμε αυτά που μας έλεγε η Επιτροπή, η γυναίκα μου θα με είχε χωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Βερένα Ρος, εκτελεστική διευθύντρια της ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους και για την πρόσκλησή σας και τη δυνατότητα να πάρω μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρίως τους κοιόδης συγητές και φυσικά τον κύριο Τόρβαλτς για την υποστήριξή τους στο θέμα του προϋπολογισμού. Όπως είπαν και οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι, είμαστε μια νέα υπηρεσία, μια νέα αρχή Έχουμε δημιουργηθεί το 2011 και δημιουργηθήκαμε επί τη βάση της σταδιακής αύξησης των πόρων μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε την αύξηση των αρμοδιοτήτων που μας έχουν δώσει οι συνομοθέτες τα τελευταία χρόνια. Έχει σημασία λοιπόν να συνεχίσουμε αυτήν την ενίσχυση έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή. Οι δημοσιονομικές προτάσεις που κάνουμε εμείς για το 2015 ανταποκρίνονται στα ελάχιστα επίπεδα τα οποία είναι απαραίτητα για να φέρουμε εις πέρας τις αποστολές που μας έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια και στον τομέα της άμεσης εποπτείας και σε σχέση με το ενιαίο εγχειρίδιο και με την εποπτεία, ε, τη σύγκληση μάλλον στις διαφορετικές ε, μορφές και πηγές εποπτείας. Ο προϋπολογισμός που έχουμε καθορίσει λοιπόν στην ΕΣΜΑ βασίζεται σε μια μηδενική βάση. Βλέπουμε εμείς πού μπορούμε να τοποθετήσουμε το προσωπικό, πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε διαδικασίες και να τις κλείσουμε ανάλογα με την επίδοση του προσωπικού και ταυτόχρονα να βάλουμε μια σωστή προτεραιότητα στις ανάγκες μας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Συνειδητοποιούμε τα δημοσιονομικά προβλήματα και την οικονομική κατάσταση και τις δυσκολίες που υπάρχουν όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο γιατί οι χώρες μέλη είναι αυτές οι οποίες δίνουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό μας. Εμείς λοιπόν με τη συμφωνία της, του Συμβουλίου Εποπτών προτείναμε μια ουσιαστική μείωση των πιστώσεων, των νέων πιστώσεων από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 γιατί συνειδητοποιούμε ε, τις δημοσιονομικές πιέσεις γενικότερα. Αλλά ταυτόχρονα ζητήσαμε και μία αύξηση στο προσωπικό η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τα τέλη από πλευράς ε, των συναλλασσομένων και των υπηρεσιών εταιριών αξιολόγησης. Οι προτάσεις λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προβληματικές γιατί αυξάνουν τις μειώσεις ακόμα περισσότερο από τις λιγότερο υψηλές που είχαμε εμείς προτείνει και δεσμεύουν και τις δυνατότητες μεγαλύτερης συνεισφοράς από τις εθνικές αρχές. 15% δηλαδή χαμηλότερες από τις προτάσεις που προτείναμε εμείς για το 2015. Είναι σοβαρό το θέμα για μια υπηρεσία η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης. Αν υποστούμε αυτές τις ε, μειώσεις ε, θα πρέπει να επανέλθουμε στις ε, προτεραιότητες των ευθυνών μας και θα αναβάλουμε και πιθανώς να ακυρώσουμε συγκεκριμένες αποστολές ιδιαίτερα στον τομέα της εφαρμογής και των πληροφορικών προγραμμάτων που θα μας δώσουν στοιχεία για να καταστεί η διαδικασία αυτή του ενιαίου εγχειριδίου λειτουργική. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να πιέσουμε έτσι ώστε να επανέλθουμε στις προτάσεις τις οποίες είχαμε καταλήξει σαν Συμβούλιο Εποπτών. Είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον Άντωνη Ντέμψη, σας ευχαριστώ. Να σας πω καταρχήν ότι εμείς στην Κομισιόν και ιδίω στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Αγορών, Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ για την πίεση στις εποπτικές αρχές να δώσουν τα αποτελέσματα που προσδοκούνται από αυτές και φυσικά αυτό σημαίνει πρέπει να έχουν τους απαραίτητους πόρους. ο κύριος Μοντάλβο από την ΕΙΟΠΑ έχει εξηγήσει τη διαδικασία που λαμβάνει η χώρα στους φορείς αυτούς και εμείς στην Κομισιόν κάθε χρόνο όπως είναι γνωστό κάνουμε την εξέταση των αιτήσεων από τους αποκεντρωμένους φορείς, τους εξετάζουμε, τους συζητούμε στους κόλπους της Κομισιόν και τελικά η Κομισιόν κάνει μια επίσημη πρόταση στις αρχές του, στην αρχή του προϋπολογισμού. και μέσα στην συζήτηση αυτή συμπεριλαμβάνεται πάντα και το θέμα των πρόσθετων εγχειρημάτων πρέπει να αναλάβουν αυτοί οι φορείς και φυσικά λαμβάνει υπόψη και το γενικό πλαίσιο της, ε, των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών προοπτικών. Το αποτέλεσμα είναι η πρόταση που είναι τώρα ενώπιον της αρχής του προπολογισμού για τους αποκεντρωμένους αυτούς φορείς, τους εποπτικούς και μπορούμε να σας παραπέμψουμε στην ανακοίνωση της Κομισιόν τον Ιούνιο του 2013 σε ό,τι αφορά το μεσοπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο και η πρότασή μας για το 2015 είναι απόλυτα σύμμορφη με αυτή την ανακοίνωση. Θα θυμόσαστε ότι για τον προϋπολογισμό του 2014 η αρχή του προϋπολογισμού είχε δώσει περισσότερα χρήματα, ένα υψηλότερο προϋπολογισμό από ότι στην αρχή είχε προβλεφθεί <clears throat> και έδωσε και πρόσθετο προσωπικό όπως είχε σχεδιαστεί για το 2015 από την Κομισιόν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο με αφήνουμε σταθερό το προσωπικό στους φορείς αυτούς, γιατί ήδη το προσωπικό που προβλεπόταν να υπάρχει το 2015 είχε εγκριθεί το 2014 και η Κομισιόν βασιστής θέση του, 2013 παραμένει στο πλαίσιο για την εξέλιξη του οργανογράμματος και γι' αυτό θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει πρόσθετο προσωπικό για το 2015. Αλλά μου υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο όμως και αυτό αναφέρθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τίθεται το θέμα της μεθόδου χρηματοδότησης αυτών των εποπτικών φορέων. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν έχει προετοιμάσει μια αναθεώρηση για το, τη λειτουργία των φορέων αυτών, όπως ζητά ο κανονισμός λειτουργίας τους, που θα δημοσιευτεί στο τέλος του μηνός. Και θα υπάρχει μέσα στην ε, επισκόψη αυτή και μια αίτηση για να εξεταστούν Όλε οι επιλογέ σε μελλοντική χρηματοδότηση των φορέων αυτών, λαμβάνοντα υπόψη και τη δυνατότητα να, καλύπτονται, να καλύπτεται μέρος ή όλο το κόστος του τους από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στην περίπτωση της ΕΣΜΑ της Αρχής για τις Αγορές υπάρχει ήδη κάποια τέτοια χρηματοδότηση. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις δυνατότητες αν υπάρχουν να μειώσουμε, να εξαλείψουμε και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών ή δυνατών. Θα είναι όμως σημαντικό να σκεφτούμε και κατά πόσο θα ήταν κατάλληλο να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα οι, τομείς, οι φορείς αυτοί που έχουν σημαντικό ρυθμιστικό καθήκον. Αλλά σίγουρα στην επισκόψη αυτή θα υπάρξει μια πιο ενδελεχής εξέταση για τα θέματα αυτά της μακροχρόνιας χρηματοδότησης αυτών των φορέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάρα πολύ σύντομα ξαναδίνω το λόγο στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Βέβαια από η δική μου άποψη βρίσκει ότι μπορεί να υπάρξει μια κάποια λύση και νομίζω ότι συμφωνούν μαζί μου και οι σκιώδεις εισηγητές. Δεν περιμένω προβλήματα. Εγώ προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα νέο σύστημα από το 17. Αυτό το κάνω για να προσφέρω υλικό για συζήτηση. Κάποιοι διαφωνούν βέβαια με αυτή την πρόταση, αλλά αυτό δεν είναι ε, ασυνήθιστο. Πρέπει να βρούμε μια λύση λοιπόν μαζί με τους κοιόδης και νομίζω ότι έχουμε κάποια θέματα τα οποία είναι περισσότερο φιλοσοφικού χαρακτήρα. Ε, λόγω του χρονοδιαγράμματος που έχουμε στην παρούσα φάση δεν θα τα λύσουμε όλα τώρα. Ευχαριστώ η προθεσμία. Είναι η 29η Ιουλίου. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει την 3η Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα θα γίνει και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Σας ευχαριστώ όλους. Η επόμενη συνάντησή μας είναι την 3η Σεπτεμβρίου. Σας εύχομαι λοιπόν καλές διακοπές.